8.30 αύριο το πρωί. Αυτή την εβδομάδα σύμφωνα με το άρθρο <clears throat> ε, του κανονισμού έχουμε προσυπογράψει με το Συμβούλιο συγκεκριμένες προτάσεις που έχουν εγκριθεί. Οι τίτλοι αυτών των νομικών πράξεων θα εμφαίνονται στα πρακτικά των, ε, της σημερινής μας συνεδρίασης. Κύριε Ντίες Δεμέρα, έχετε ζητήσει να παρέμβετε. Έχετε τον λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ανεκτικότητά σας. Θέλω να αναφερθώ σύντομα Πρόεδρε στα θύματα. Τα θύματα που ήταν... Ε,